έλαβα από το ΕΛΚ ε, ένα αίτημα ε, σχετικά με τις αντιπροσωπίες ε, και τον διορισμό συναδέλφων. Έχει δοθεί ο κατάλογος, αν υπάρχουν αντιρρήσεις θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται.